Καλησπέρα. Ξεκινά η συνεδρίασή μας. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης ε, είναι ένα θέμα το οποίο μπορείτε τώρα να μας πείτε αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια, όχι. Άρα εγκρίνεται.